Ούτε λεπτό παραπάνω. To, to open the meeting. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Πρόκειται για κοινή συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών ε, Υποθέσεων. Δεν είναι εδώ ο κύριος Βόμπεντ. Έχουμε τη Μάντι Ντελβό που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γιούρη και θα συμπροεδρεύει μαζί μου. Ε, ολοκληρώσαμε το έργο της Ομάδας Εργασίας για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία και τώρα περνάμε, ελπίζουμε, στο τελευταίο στάδιο αυτής της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για την ε, ε, σωστή εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας. Σήμερα έχουμε την πρώτη συνάντηση η οποία θα αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα των συζητήσεων για την έκθεση. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν δύο συνεισηγητές, ο Ρίτσαρ Κόρμπετ που εκπροσωπεί την Επιτροπή ΑΦΚΟ και ο άλλος είναι ο Πάβελ Σφόμποντα ο οποίος ε, εκπροσωπεί την Επιτροπή Γιούρι. Ε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν να δώσω το λόγο στο Ρίτσαρτ για να μας πει ότι θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε αυτό το στάδιο των εργασιών. Ωραία λοιπόν. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε από αυτά που είχαμε τις διάφορες πτυχές ε, της Διοργανικής Συμφωνίας ε, που εγκρίθηκε το Μάρτιο πέρσι, το Μάρτιο του 2016, για να δούμε πώς προχωρούσε η εφαρμογή. Είναι βέβαια η αρχή ακόμα από πολλές ε, ε, πλευρές και υπάρχουν δύο εκκρεμότητες ε, τα οποία, οι οποίες ακόμα απαιτούν διοργανική συμφωνία. Το θέμα του χαρακτηρισμού και της διαφοροποίησης μεταξύ εκτελεστικών πράξεων και πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Ο υποφαινόμενος και ο συνάδελφος είναι αρμόδιοι για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των οργάνων και οι διαπραγματεύσει που μπορεί να οδηγήσουν σε διεθνεί συμφωνίε ε, του κυρίου Μπροκ και Λάγκε που είναι οι διαπραγματευτέ του Κοινοβουλίου. Δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτέ οι διαπραγματεύσει ακόμα, είναι σε εξέλιξη. Επομένω, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε ακόμα αυτέ τι πτυχέ. Απλώ ε, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία. Η ομάδα εργασία, βέβαια, ε, εξέτασε τι διάφορε πτυχέ, τι οποίε έχει υπάρξει μια αρχική συμφωνία. Διοικητικές αλλαγέ. Το Κοινοβούλιο μέσω της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει πλέον 7 ε, τμήματα στην υπηρεσία που ασχολούνται ε, με αξιολογήσει αντικτύπου, είτε αξιολόγηση των αξιολογήσεων αντικτύπου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν το ζητούν οι επιτροπές. Εξετάσαμε τις αλλαγές στον κανονισμό του Κοινοβουλίου που εφαρμόστηκε μετά από την έκθεσή μου για τη γενικότερη αναθεώρηση του κανονισμού πέρσι. Ε, με σκοπό να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ε, ανατίθεται εντολή ε, σε όσους συμμετέχουν στις τριμερείς διαπραγματεύσεις από πλευράς ε, Κοινοβουλίου για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος ε, για το κατά πόσον θα δίνεται ή δεν θα δίνεται τελικά η εντολή. Αποφασίζει το Κοινοβούλιο. Εξετάσαμε πώς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει και το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Ελέγχου που αντικαθιστά το προηγούμενο ε, Συμβούλιο Αξιολόγησης και την ανεξαρτησία των μελών του Συμβουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάσαμε πώς εξελίσσεται αυτό. Ακόμα είναι πολύ νωρίς βεβαίως για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ε, πρέπει να δούμε τις προκλήσεις. Εξετάσαμε το REFIT, το πρόγραμμα για το πώς προχωρά το REFIT. Ε, δεν έχουμε ακόμα εξετάσει, αλλά ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, κάνει την πρώτη ε, διεθνή έρευνα για την επιβάρυνση στις μικρές επιχειρήσεις, την οποία λάβαμε μόλις τον περασμένο μήνα εδώ στο Κοινοβούλιο. Επομένως, ακόμα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα αυτή τη στιγμή για το πόσο καλά λειτουργεί αυτό, όταν ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση του Κοινοβουλίου για την πρώτη έρευνα. Ε, εξετάσαμε το θέμα της ε, υπερβολικής νομοθεσίας από πλευράς κρατών μελών, το gold plating, ε, είδαμε τον προγραμματισμό, τι διαδικασίες έχουμε εκεί ε, και προχωρούν ακόμα οι εργασίες. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος για τη βάση δεδομένων μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πολλά πράγματα λοιπόν είναι σε εξέλιξη σε διάφορα επίπεδα και με αρκετούς που είναι αρμόδιοι για τα θέματα αυτά, εξού και για το, αυτό το λόγο και η ομάδα εργασία για να δούμε ε, ο ένα να κοιτάει από τη μια, ο άλλο από την άλλη και να συντονίζουμε πώ γίνονται όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό όσον αφορά το ψήφισμα ή την έκθεση που πρέπει τώρα να εξετάσουμε. Όπως είπα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ακόμα νωρίς για κάτι τέτοιο ε, υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα συμφωνημένο, επομένως πρέπει να γίνει μια πρώτη προσπάθεια να ε, σημειώσουμε τι συνέβη, να ενθαρρύνουμε συμφωνία στις δύο εκκρεμότητες που έχουμε, ε, στις οποίες ακόμα η διοργανική συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί και να δούμε κατά πόσον η εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας θα μπορούσε να βελτιωθεί. Όπως είπα, είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά ε, οι συνάδελφοι μπορεί να έχουν κάποιες ιδέες από αυτόν. Αυτό το οποίο δεν θα ήθελα να συμβεί είναι να ξεκινήσει ε, τώρα μια προσπάθεια να ξανανοίξει η διοργανική συμφωνία πέρσι την υπογράψαμε. Επομένως το πρώτο στοιχείο είναι να την εφαρμόσουμε σωστά, να είμαστε βέβαιοι ότι εφαρμόζεται πλήρως και ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει τα εκμεταλλευόμαστε δεόντως πριν προχωρήσουμε στην πρόταση να γίνει νέα διαπραγμάτευση ή να ξαναγραφτεί από την αρχή. Δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό σε αυτή τη φάση. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του επόμενου κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, Ρίτσαρτ. Ο Άξελ θα διαβάσει τη δήλωση του κυρίου Σβόμποντα. Οπότε έχεις δύο τους οποίους πρέπει να αντικαταστήσεις. Εκ μέρους λοιπόν του συναδέλφου κυρίου Σφόμποτα έχουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις γιατί στις 7 Δεκεμβρίου ε, θα λάβετε και το περιεχόμενο της ε, μελλοντική του έκθεσης. Ο κύριος Φόμποτα θα θέλει να ευχαριστήσει όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας και τους εμπειρογνώμονες για τη συμμετοχή τους όπως επίσης να μας πει πως η ομάδα εργασίας που στάθηκε το Μάιο του 2016 έκανε νέα συνεδριάσεις με πλήρη ανταλλαγή απόψεων, πολύ καρποφόρα, με μέλη από άλλες επιτροπές και με εκπροσώπους ε, άλλων επιτροπών, άλλων υπηρεσιών ε, με τρόπο ιδιαίτερα ικανοποιητικό, μια και η συνεισφορά ε, όλων στην ε, ομάδα εργασίας ε, έφερε πολλά θετικά για τη μελλοντικό σχέδιο έκθεσης αυτό της Επιτροπής Γιούρη και της Επιτροπής ΑΦΚΟ για την εφαρμογή της νομοθεσίας εδώ, κυρίως στο θέμα του πολιετούς προγραμματισμού και αυτό στα πλαίσια της κοινοβουλευτική εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει, καλύτερη νομοθέτηση και τα σχετικά εργολεία, όπως επίσης ε, το θέμα της συλλογικής μελέτης, τα νομοθετικά εργαλεία, η επιλογή νομικής βάσης, οι εφαρμοστικές και κατεξουσιοδότηση πράξεις και κυρίως το κριτήριο ε, διαχωρισμού, η διαφάνεια και ο συντονισμός της νομοθετικής διαδικασίας, η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, η απλούστευση και κυρίως ε, η έρευνα για το ετήσιο βάρος. Ο κύριος Φόβοντα με προσδοκία αντιμετωπίζει τη συνεργασία με τον κύριο Κόρμπετ και με τους συναδέλφους από όλες τις επιτροπές που θα συνεισφέρουν στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ Άξελ. Ποιος ήταν ο επόμενος ομιλητής. Βλέπω είναι και άλλοι. Δύο λοιπόν συνάδελφοι. Ο κύριος Μάρκος Πίτερ πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα μιλήσω γερμανικά. Όλα καλά λοιπόν. Εφαρμόζουμε διοργανική συμφωνία. Ακούμε ότι η νομική υπηρεσία έχει διαβουλευτεί. Ακούμε από τον εισηγητή ότι δεν ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες ε, δυνατότητες πρωτού εξαντλήσουμε τις δυνατότητες ε, της παλιάς. Κύριε Κόρπετ, έχετε δίκιο, αλλά δεν εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Αντιθέτως, τις μπλοκάρουμε. Υπάρχει τμήμα για μελέτες αντικτύπου εντό του Κοινοβουλίου. Εφτά φορές από τότε που υπάρχει αυτό το τμήμα, Ε, την έχουμε εκμεταλλευτεί και αυτό είναι αποτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, η Επιτροπή μας ε, το έχει ζητήσει επανειλημμένα, αλλά θα πρέπει η πλειοψηφία των συντονιστών θα πρέπει να συμφωνήσει για κάτι τέτοιο, κάτι που ουσιαστικά ποτέ δεν γίνεται. Έχουμε υποβάλει το θέμα αυτό στους πρόεδρους των επιτροπών. Τέσσερις ε, πρόεδροι των επιτροπών θέλουν να μειώσουν το κατόφλι. Δύο συντονιστές ε, να συμφωνούν, για παράδειγμα, ή ο εισηγητής ε, και ένας ή δύο συντονιστές. Να υπάρχει χαμηλότερο κατόφλι για τη χρήση αυτής της δυνατότητας, αλλά αυτό έχει μπλοκαριστεί πολιτικά από την ΑΦΚΟ και άλλες επιτροπές και έτσι τελικά δεν ε, έχει περάσει το θέμα. Γι' αυτό εγώ σιγά σιγά εγκαταλείπω τα όπλα. Διότι ε, μπλοκαριζόμαστε πολιτικά κάθε φορά. Δεν έχω και πια διάθεση να συμμετέχω στις συναντήσεις που ανέφερε ο Αξελφός. Ε, δεν γίνεται τίποτα, ούτε συζητιέται τίποτα, ούτε αποφασίζεται τίποτα ένας ευρωβουλευτής σε δύο να ήταν παρόντες κάθε φορά. Ε, θα πρέπει νομίζω να είμαστε ειλικρινεί σχετικά με το τι γίνεται στο Κοινοβούλιο. Τίποτα δεν γίνεται. Και θα πρέπει να ασκήσουμε αυτοκριτική και να πούμε ότι αν ε, τόσο πρόχειρα αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε καθόλου. Και μια τελευταία ε, παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει όλη την καλή βούληση. Αυτό δεν το ανέφεραν ε, οι δύο συνάδελφοι. Υπάρχει πρόσφατα Δημιουργήθηκε πρόσφατα μια task force για την επικουρικότητα που δημιούργησε ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ. Έχουμε λοιπόν πάλι άλλη μια νέα δομή ε, για την εποπτεία της κατάστασης ε, και ε, το χειρότερο καλέσαμε αυτό το Συμβούλιο Ελέγχου, το Scrutiny Board, στην Ήτρε, η οποία όμως, το, το οποίο όμως αυτό το Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Μόνο νέου τίτλου στι εφημερίδε είχαμε και λυπάμαι πάρα πολύ που είμαι τόσο αρνητικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Προτού να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Γνωρίζετε περίπτωση επιτροπής όπου να ζητήθηκε ε, μελέτη αντικτύπου και να ε, το αρνήθηκε η επιτροπή. Δεν υπήρξε τέτοιο μπλοκάρισμα, απλά καταλήξαμε σε, στο συμπέρασμα ότι για να αλλάξει το κατόφλι θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός. Και γι' αυτό στην Επιτροπή της ΑΦΚΟ επιστήσαμε την προσοχή της ομάδας εργασίας στο θέμα αυτό. Και με το θέμα αυτό θα ασχοληθούν τώρα οι συνάδελφοι που θα ασχοληθούν και με την έκθεση αυτή. Να παρουσιάσετε λοιπόν ε, τα στοιχεία όσα έχουν. Δίνω το λόγο στη Σίλβια Κάουφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την πρόεδρο της ΑΦΚΟ που έθιξε το θέμα. Διότι ξέρω ότι το θέμα των ε, μελετών αντικτύπου ε, είναι θέμα που συζητιέται πολύ στο Κοινοβούλιο και υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ε, στο θέμα και διαφορετικές απόψεις. Εγώ πάντως ε, δεν γνωρίζω περίπτωση όπου να μην ανατέθηκε μια μελέτη αντικτύπου ενώ να το έχει ζητήσει η αρμόδια επιτροπή. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού. Τώρα όμως που μιλάμε για το θέμα αυτό θα ήθελα να μην αναφερθώ σε ένα σωρό άλλα θέματα, να πω απλά στον Ρίτσαρτ Κόρμπετ ότι συμφωνώ με αυτά που είπε, ότι δεν είναι δυνατόν να αμφισβητήσουμε αυτή τη στιγμή την διοργανική συμφωνία και να ζητήσουμε τροποποιήσεις. Όσον αφορά την μελέτη αντικτύπου και το, το Συμβούλιο Ελέγχου, το Scrutiny Board, θα ήθελα να πω το εξή. Ε, η ομάδα αυτή δεν ε, υποβάλλει προτάσεις ε, δεσμευτικές. Ε, άλλωστε δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει την νομοθετική διαδικασία. Αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Ο συνάδελφος Πίπερ παραπονιέται ότι ε, το Συμβούλιο Ελέγχου δεν έχει ακολουθήσει επιθυμία της ε, Επιτροπής. Αλλά εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη σελίδα 3 της έκθεσης, όπου λέει ότι το Συμβούλιο Ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και, διαβάζω στα αγγλικά, τα μέλη του ε, δεν υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο. Και εγώ σκόνταψα στο θέμα αυτό κατά την ανάγνωση της έκθεσης ε, από τη μία ε, ανεξαρτησία, αυτονομία, αλλά από την άλλη ε, έχουμε τρεις εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία τέτοια ομάδα εκτός οποιοδήποτε πολιτικού ελέγχου. Νομίζω ότι οι συγητές θα πρέπει να προσέξουν το θέμα αυτό. διότι δεν μπορούμε να έχουμε μια τόσο αυτόνομη επιτροπή. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Και εναπόκειται στους εισηγητές να χειριστούν το θέμα ώστε να, βρουν, να συγκεντρώσουν όσο γίνεται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Μια τελευταία παρατήρηση. Δεν ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό, αλλά <laughs> με προκαλεί ο συνάδελφος Πίπερ. Όσον αφορά αυτήν την ειδική ομάδα για τα θέματα επικουρικότητας, ε, έχει νομίζω άλλους στόχους. Ε, καλό είναι ότι δημιουργήθηκε, καλό είναι ότι εκπροσωπείται το Κοινοβούλιο. Ε, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη το θέμα της επικουρικότητας, ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά το να τα μπερδέψουμε όλα αυτά μεταξύ τους ε, δεν βοηθάει κανέναν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σίλβια. Να δώσω το λόγο στον Σαγιάτ Καρίμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε που έφτασα καθυστερημένα. Η παρουσίαση έγινε λίγο πριν μπω στην ε, αίθουσα. Έχω πρόβλημα με το μικρόφωνο μας, μετακινηθώ δίπλα. Ah, Έχω δύο-τρεις πολύ σύντομες ε, παρατηρήσεις. Καταρχήν με εντυπωσίασαν τα σχόλια και με παραξένευσαν τα σχόλια που άκουσα πως το κοινοβούλιο μας δεν θεωρείται από πολλούς να έχει κάνει πολλά τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Μα νομίζω ότι η απόδειξη που καταρρύπτει αυτή την άποψη είναι αυτό που είδαμε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί θα δείτε πως εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο κείμενο που είναι copy-paste των όσων προτείναμε εμείς τις σχετικές αναφορές από τις σχετικές επιτροπές τούτου του Κοινοβουλίου και ο αντιπρόεδρος κύριο Τίμερσμαντ τα συμπεριέλαβε ως κομμάτι της μεταρρυθμικής του προσπάθειας. Οπότε τέτοιου είδους επιχειρήματα κασταρρύπτονται εύκολα. Ρίτσαρντ, μπορεί να σε πέτυχα στο τέλος, αλλά και κάνω λάθος ίσως. Αλλά η εντύπωση που μου δημιουργείται είναι ότι είπες ότι θα ήταν καλύτερα να παγιώσουμε τη θέση μας και να μην προχωρήσουμε περαιτέρω ε, το θεματολόγιο αυτή τη στιγμή. Αν σε παρανόησα, λυπάμαι πολύ. Αλλά αν αυτό ζητά, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε όσο δυνατόν πιο φιλόδοξοι από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί υπερβολικά πολλοί από τους συμπολίτε μας έχουν την εντύπωση για τη δική μας νομοθετική ε, διαδικασία εδώ, ε, η οποία πραγματικά πόρο απέχει από την πραγματικότητα και για τα εθνικά κοινοβούλια μέχρι επίσης μέσω των δικών μας διαδικασιών εδώ ε, συμπεριλάβουμε, συμπεριλάβουμε στην ε, δράση μας όσο το δυνατόν πιο στενά τα εθνικά κοινοβούλια έτσι ώστε να έχουν αυτά την ευθύνη για τις τελικές ε, αποφάσεις θα είμαστε πάντα στην περίπτωση της Ευρώπης Αλακάρτ, όπου τα όπου τα κράτη-μέλη όταν οι κυβερνήσεις βλέπουν ότι έχουμε λάβει ένα μέτρο δημοφιλές λέει πως το προώθησαν οι ίδιες και όταν κάτι δεν είναι δημοφιλές το ρίχνουν στην Ευρώπη και οι πολίτες μας δεν γνωρίζουν πως λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες, τι έχει συμβεί και αυτό είναι κάτι που εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να το αντιμετωπίσουμε και να αναλάβουμε εμείς τον ηγετικό ρόλο γιατί εδώ σε διαδικαστικό επίπεδο δεν είμαστε πάντα συστηματικοί ε, που εμείς ως συνάδελφοι επιλέγουμε τις εναλλακτικέ που είναι διαθέσιμες. Με τις επιπτωσιολογικές μελέτες, για παράδειγμα, έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι να ελέγχουμε κατά πόσο οι επιτσολικέ μελέτες τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι σωστές όταν προσκομίζονται και δεύτερον με τις δικέ μας, με δική μας πρωτοβουλία. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να τις έχουμε στα τέλη, για παράδειγμα, διαδικασία τριμερού διαλόγου και όχι στην αρχή αυτού και μπορεί να γίνουν κάποιες ουσιαστικές αλλαγές. Και πάλι συγγνώμη αν τα σχόλιά μου δεν είναι απολύτως σωστά, γιατί κάποιες από τις παρουσιάσεις έλαβαν χώρα πριν μπω στην αίθουσα. Αλλά ήθελα να τα πω για να γραφτούν κάπου στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα λεπτά μας μένουν. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Ή αν μπορώ να δώσω το λόγο στο Ρίτσαρντ. Ρίτσαρντ, έχει το λόγο. Για να κλείσουμε. Και αν χάσουμε τη διερμηνία, λυπάμαι πολύ, οι διερμηνοί σε τέσσερα λεπτά μπορούν να φύγουν. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσω του κυρίου Βος και τον κύριο Σφόποντα. Λυπάμαι πολύ που δεν ήταν εδώ. Και σας ευχαριστώ πολύ και προς το προσωπικό που δεν το είπα προηγουμένως. Δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά για το θέμα. Πιστεύω πως, όπως είπε και η κυρία Κάφμαν, είναι θέμα σωστής ισορροπίας που πρέπει να πετύχουμε. Και όταν ακούω σχόλια που λένε πως δεν έχει γίνει τίποτα, δεν καταλαβαίνω πως αυτό είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση ε, γιατί πολλά έγιναν και δεν μπορούμε να τα αγνοούμε λέγοντας πως δεν πως δεν έγινε τίποτα. Άλλαξαν οι κανόνες, άλλαξαν οι διαδικασίες. Δεν είναι δίκαιο να λέμε πως δεν έγινε τίποτα ίσως δεν παρκή. Ίσως θα πρέπει να γίνει καλύτερα. Αλλά το να πει κανείς πως δεν έχει γίνει τίποτα είναι πραγματικά πολύ απορριπτικό για την όλη διαδικασία. Και οδηγούμε τώρα στα σχόλια του κυρίου Καρίμ για το τι κάνουμε με την έκθεση αυτή. Η διαφοροποίηση που έχει λάβει χώρα για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και για το κατά πόσο μπορούν να πάνε καλύτερα τα πράγματα, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Δεν, Δεν ξέρω τι εννοείται, αναθεώρηση ή επαναδιαπραγμάτευση. Γιατί εγώ αυτό που θα έλεγα είναι το εξή. Μόνο ούτε χρόνος δεν έχει περάσει, ανάμιση χρόνος πέρσι το Μάρτιο. Ε, πετύχαμε την, διαθέσιμη, την συμφωνία μεταξύ θεσμών. So Και δεν νομίζω πως είναι ο χρόνος τώρα να κάνουμε αλλαγές σε αυτή τη διαθεσμική, διοργανική με συμφωνία και θα πρέπει να δούμε ζητήματα σαν αυτά που έθεσε ο συνάδελφος. Είναι δύσκολο για τι άλλε επιτροπέ, να λαμβάνουν επιτοσιολογικές μελέτες για να δούνε τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχω ακούσει να έχουν αρνηθεί αυτό το δικαίωμα σε κάποια επιτροπή. Πάντως θα τα δούμε. Και μια τελευταία παρατήρηση για το νέο αυτό σώμα, για την επικουρικότητα, τα όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Δεν ξέρω πόσο αυτό έχει συνέπειες για τα όσα εμείς κάνουμε για την καλύτερη νομοθεσία. Μιλάμε για καλύτερη νομοθεσία, better regulation, όχι απορρίθμιση, deregulation και θα με έχετε ακούσει να το λέω αυτό στο παρελθόν. Η ιδέα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετεί υπερβολικά πολύ σε θέματα τα οποία δεν επιθυμούν τα κράτη-μέλη είναι υπερβολή. Καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί να συμφωνηθεί εάν δεν εγκριθεί όχι μόνο από εμάς που είμαστε ιερετοί, αλλά και από το Συμβούλιο. Και ποιο βρίσκεται στο Συμβούλιο, οι Εθνικοί Υπουργοί. Υπουργοί που εκπροσωπούν εθνικές κυβερνήσει, λογοδοτούν σε εθνικά κοινοβούλια. Και πολλές φορές μπορεί να ζητούν από του υπουργού του να λογοδοτούν, αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την παραμικρή τάση να ε, τα λύνουν όλα κεντρικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί έτσι ε, ε, δεν γίνεται. Επίσης πολλές φορές χρειάζεται ομοφωνία, πολλές φορές ειδική πλειοψηφία. Οπότε δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν εχέγγυα στη δική μας νομοθετική διαδικασία έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι πως τα κράτη-μέλη δεν χρειάζεται να δεχτούν νομοθεσία την οποία δεν επιθυμούν. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία κάθε φορά ε, υπέρ της ανάγκης να νομοθετήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ρίτσαρτ, σας ευχαριστώ όλους και πριν φύγουμε να σας ενημερώσω πως θα γίνει μία συνάντηση των δύο επιτροπών στις 7 Δεκεμβρίου 9 με 9 και 45 στα πλαίσια του χρόνου που έχει η Επιτροπή Γιούρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Dear colleagues, just if there is anybody from AFCO assistance here, we are having extraordinary meeting, I am told, on 11th for the vote